Η κυρία Μογκερίνη θα λάβει τώρα τον λόγο. Παρακαλώ. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. I know how the is after a vote. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ολομέλεια μετά την ψηφοφορία. Συζητήσαμε το θέμα της ισιας, στο περιθώριο σε εισαγωγικά το βάζω, της συνάντησης. Είπαμε ότι η Λιβύη είναι ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη νότια γειτονία. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τις γειτονικές χώρες, ξεκινώντας από την Τινησία. Και λίγες μέρες μετά, δυστυχώς, συζητάμε για μια πολύ ευαίσθητη πλέον κατάσταση μετά την επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας. Η Τινησία είναι μια ειδική χώρα γείτονα για μας. Είναι μια χώρα που δείχνει ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμοί στη δημοκρατία και η δημοκρατία μπορεί να είναι το μέλλον της περιοχής. Εγώ εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ένα νέο παιδί που πήρε μέρος μετά την απόπειρα στην Τινίδα και είπε ότι αυτοί που τρομοκρατούν, που ε, τους τρομοκράτες είμαστε εμείς, δηλαδή η μελλοντική γενιά των νέων τηνησίων. Η μοναδική καλή απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε είναι να στηρίξουμε το παιδί αυτό, να στηρίξουμε αυτό το αγόρι και αυτά τα κορίτσια που είχαν κατέβει σε διαδηλώσεις αντιδρώντας την επίθεση όπως και οι Γάλλοι πολίτες είχαν αντιδράσει στις επιθέσεις του Ιανουαρίου στο Παρίσι. Όλοι οι Τινήσοι, ιδιαίτερα οι νέες γενιές, πιστεύουν στο μέλλον μιας ελεύθερης δημοκρατικής χώρας. Την παραμονή της επίθεσης, εμείς εδώ συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών για το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τινησία. Από τη μία συζητούσαμε όπως συζητάμε συνήθως τέτοιες, τέτοιες ε, ευκαιρίες για τις εξελίξεις στη χώρα τον τελευταίο χρόνο, την υιοθέτηση ενός νέου συντάγματος, τις προεδρικές εκλογές, μια κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά συζητήσαμε και τα θέματα που καθιστούν την χώρα αυτή ε, εύθραυστη η νεολαία της χώρας αυτής, η οποία είναι πολύ υψηλά εκπαιδευμένη, αλλά όμως έχει τεράστια ποσοστά ανεργίας. Αναζητούν θέσεις στην κοινωνία οι νέοι και κυρίως οι νέες στην Τινησία. Υπάρχουν ε, πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα σε επίπεδο δημοκρατικής ε, διαδικασίας και αναφέρομαι στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν στο τέλος του χρόνου. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα της χώρας. Υπάρχουν περιοχές με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους σε επίπεδο εισοδημάτων, σε επίπεδο κοινωνικό, διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Συζητήσαμε επίσης και την δυνατότητα αδελφοποίησης ορισμένων περιοχών και πόλεων στην Τινησία με αντίστοιχες περιοχές και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και θέμα επίσης ασφάλειας για τη χώρα. Υπάρχουν απειλές από την ε, μία χώρα ε, στην οποία Υπάρχουν προβλήματα με τους πρόσφυγες, υπάρχει θέμα ελέγχου των συνόρων Ε, είπαμε ότι θα υπογράψουμε και συμφωνίες συνεργασίας έτσι ώστε να ανοίξουμε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα προς την ισίους νέους την νησίων, την ισιακές επιχειρήσεις, ερευνητές, καθηγητές που θέλουν να πάρουν μέρος στα ευρωπαϊκά προγράμματα με πιο δεκτικό τρόπο. Έτσι θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και θα υπάρξει μια επίσκεψη υψηλού επίπεδου μετά από τη δική μου επίσκεψη στην Τίνιδα. Εγώ είχα πάει εκεί τον μήνα Φεβρουάριο, μια εβδομάδα μετά από τον σχηματισμό της καινούργια κυβέρνησης και την επόμενη Τρίτη μαζί με τον πρόεδρο Τούσκ θα επισκεφθούμε τη χώρα. Την ημέρα μετά την επίθεση μίλησα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της χώρας ανταλλάξαμε συλληπιτήρια. Εγώ μίλησα για τα θύματα της, ε, των τινησίων, μάλλον τους τινήσιους που έπεσαν θύματα της απόπειρας και αυτός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο, την απώλεια ζωής Ευρωπαίων πολιτών. Μου είπε λοιπόν ένα πράγμα ο προτιμήσιος Πρωθυπουργό ότι, μπορούμε, ε, ότι κάνουμε μάλλον ό,τι μπορούμε έτσι ώστε τέτοιου είδους επιθέσεις να μην διακόψουν τις διαδικασίες μας οι οποίες είναι διαδικασίες εύθραστες και είπε ότι εμείς βλέπουμε την Ευρώπη σαν την καλύτερη μας φίλη. Πέρασα το μήνυμα Ξεκινήσαμε τη συνάντηση του, Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών με ενός λεπτού σιγή και προσπαθήσαμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε πράγματι φίλοι ε, με τους τινήσιους σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Θα πρέπει να αυξήσουμε την συνεργασία μας μαζί τους σε τέσσερα επίπεδα μπορεί να γίνει αυτό, στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της ε, δημοσιονομικής υποστήριξης και στον τομέα των περιφερειακών σε σχέση με τη Λιβύη. Να σταθώ τώρα ξεχωριστά σε αυτά τα θέματα. Πρώτον, στον τομέα της ασφάλειας. Είναι προφανές ότι η ασφάλεια βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας και του δημοκρατικού συστήματος. Ισχύει και το αντίστροφο όμως. Μπορεί να υπάρξει ασφάλεια με γνήσιες δημοκρατικές δομές, σε ε, του δικαίου και του του κράτους δικαίου και χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει δίκαιο, δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιο. Έχουμε λοιπόν περάσει σε τρεις ε, έρευνες οι οποίες γίνονται στην την Ισία, τις οποίες ε, εμείς συμμετέχουμε. Η μία αφορά την δικαιοσύνη, η άλλη αφορά την διαχείριση των συνόρων και η τρίτη την δημόσια διοίκηση. Έχουν ξεκινήσει κάποια προγράμματα στον τομέα της, του ελέγχου των συνόρων για τη μείωση των κινδύνων και από την τρομοκρατία και θα ενισχύσουμε τις διαδικασίες με 25 εκατομμύρια ευρώ. Θα συνεργαστούμε και με τους εταίρους μας, τους τινησίους και στις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα βέβαια, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες επαχές. Ε, ο συντονιστής μας είχε πάει στην Τινίδα λίγες μέρες πριν από την επίθεση και συζήτησε με τους ομολόγους του νέα πεδία συνεργασίας, διάλογο για την τρομοκρατία και κάποια συζήτηση για πακέτα μέτρων τα οποία ελπίζω να τεθούν σε λειτουργία τις επόμενους μήνες. Η εταιρική αυτή σχέση γίνεται σε ισότιμο απολύτως επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η υποστήριξη της σταθερότητας στην Τινησία δεν απαιτεί μόνο βούληση. Απαιτεί, και το είπα αυτό και δημόσια και ιδιωτικά, υποστήριξη στην οικονομία, στην οικονομική μετάβαση και στη δημοκρατική μετάβαση. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Καταρχάς, οικονομική βοήθεια. Από το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διπλασιάσει ε, τα αρχικά ποσά για την Τινησία το 2014 170 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στην Τινησία. Η μικροχρηματοδοτική βοήθεια, γύρω στα 300 εκατομμύρια σε δάνεια, έρχεται συμπληρωματικά. Οι προβλέψεις για το 2015 δεν έχουν καθοριστεί πλήρως αλλά συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Χάν έτσι ώστε η Τινησία να πάρει αυτά τα οποία τη αξίζουν και αυτά τα οποία χρειάζεται, γιατί αυτό είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Η χρηματοδοτική βοήθεια περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να αναλυφθούν έτσι ώστε να συνοδεύσουν την χώρα αυτή στην πορεία της προς τις μεταρρυθμίσεις ενίσχυσης της δημοκρατίας και της οικονομίας. Ε, περαιτέρω ολοκλήρωση της, της ε, οικονομίας της Τινησίας στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά με τους τρόπους βέβαια που αρμόζουν και ταιριάζουν στα δικά της ε, χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα συζητά τα θέματα αυτά με τις νέες αρχές της Τινησίας από τον προηγούμενο μήνα. Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία. Είναι σημαντικό επίσης να δώσουμε κάποια θετικά μηνύματα προς τους επενδυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν την οικονομία στη χώρα. Αυτό θα αποδώσει και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βέβαια πρέπει κυρίως βραχυπρόθεσμα να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Ήδη από, τους, από τις αρχές του χρόνου εμείς έχουμε ρυθμίσει ε, τις ποσοστώσεις μας στον τομέα των εισαγωγών ελαιολάδου κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τη χώρα αυτή. Μελετάμε επίσης ε, και τη συμμετοχή της Τινησίας σε προγράμματα έρευνας. Αυτά είναι δύο παραδείγματα. Θα υπάρξουν και άλλα στο μέλλον, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα ε, και μπορούμε να βοηθήσουμε σε σημαντικό επίπεδο. Ε, εκεί όπου πρέπει να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία είναι το θέμα της Λιβύης. Από τη μία έχουμε το θέμα των συνόρων και από την άλλη έχουμε το γενικότερο πρόβλημα της Λιβύης που επηρεάζει την κατάσταση στην Τινησία. Νομίζω ότι ε, θα πείτε αρκετά και εσείς γύρω από το θέμα αυτό και γι' αυτό επιφυλάσσομαι ε, να σας ακούσω πρώτα. Αλλά πάντως είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Εμείς σε επίπεδο διπλωματίας πιέζουμε ακόμα περισσότερο εγώ η ίδια οργάνωσα μια συνάντηση 24 ε, δημάρχων από τη Λιβύη εδώ και δύο μέρες στις Βρυξέλλες ε, ακούγοντας τους ε, πραγματικά καταλαβαίνει κανείς γιατί μόνο οι δήμαρχοι μπορούν να καταλάβουν τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουν οι πολίτες. Από την άλλη είδε κανείς ποια είναι τα αισθήματα των ανθρώπων αυτών και η ανάγκη την οποία νιώθουν για να προχωρήσουμε σε μια πολιτική συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στη Λιβύη να κάνει μια νέα εκκίνηση. Μέτρα εμπιστοσύνης και μια έκκληση προς τον πολιτικό κόσμο να δώσει τα απαιτούμενα, τις απαιτούμενες λύσεις. Ξέρετε ότι ε, τίθεται το θέμα ενός νέου πολιτικού πλαισίου και στα πλαίσια των συναντήσεων στο Ραμπάτ αλλά και στα πλαίσια του Τομπρούκ, της συνάντησης του Τομπρούκ και της Τρίπολη της ε, ε, Λιβύη. Λοιπόν, ελπίζουμε αυτά όλα να διευκολύνουν και την καθημερινότητα των τινήσιων φίλων. Και πριν κλείσω ένα στοιχείο ακόμα, και αυτό αφορά τον δικό σας ρόλο και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά και η κοινοβουλευτική συνεργασία είναι αναπόσπαστο τμήμα της βοήθειας την οποία αναζητάει την Ισία. Νομίζω ότι η δική σας εμπλοκή θα έχει τεράστιες, τεράστια θετικά στοιχεία. Ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία από το 2014 στα πλαίσια της βοήθειας προς την Βουλή της Τινησίας. Αυτό είναι πολύ θετικό και για αυτούς και για μας ε, προβλέπεται η σύγκληση της Μικτής Επιτροπής, της Διακοινοβουλευτικής, γενικά ενισχύοντας ε, τους θεσμούς μας με τη νέα Βουλή της Τινησίας θα ενισχύσουμε ε, την δημοκρατία στη χώρα αυτή. Είδαμε, είδαμε στην τηλεόραση να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της χώρας κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την ώρα που γινόταν η επίθεση ήταν ένας τρόπος έτσι ώστε ε, ε, να δείξουν το τι πιστεύουν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τους βοηθήσουμε, πρέπει να τους συμπαρασταθούμε και να τους ενισχύσουμε και να τους πούμε ότι δεν θα μείνουν ποτέ μόνοι γιατί μπορούν να μας έχουν φίλους, φίλους οι οποίοι θα τους στηρίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε Μογκερίνη. Ξέχασα να αναφέρω ότι σε αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης πέρα από α, τις παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων δεν θα γίνει καστιάες. Και παρακαλώ να τηρήσουμε αυστηρά τον, τους κανονισμούς γιατί έχουμε σοβαρή καθυστέρηση. Πρέντα παρακαλώ δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη. Αμέσως μετά την τρομερή επίθεση κατά το Μουσείο του Μπάρντο, η ομάδα του ΕΛΚ καταδίκασε την πράξη αυτή. Και εγώ ίδιος πριν από μια εβδομάδα στα κοινωνικά δίκτυα υπέβαλα τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και εξέφρασα την πλήρη μας αλληλεγγύη. Η επίθεση του Μπάρντο στόχευσε την χώρα που έχει κάνει τις περισσότερες προσπάθειες για να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις της Αραβικής Άνοιξης. Πέρα από τα αθώα θύματα, έγινε η επίθεση κατά της δημοκρατικής μετάβασης της Τινησίας που είναι μοναδικό φαινόμενο στον αραβικό κόσμο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η επίθεση της Τινησίας δεν είναι μόνο κατά του εταίρου μας, αλλά και κατά ημών των ιδίων. Καταρχήν αυτό φαίνεται διότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Έπειτα διότι η ασφάλεια της Μεσογείου είναι και δική μας ασφάλεια. Και τέλος, διότι η επίθεση του Μπάρντο είναι επίθεση κατά των αξιών μας ανοχή και θεμελιώδης ελευθερίες. Το Νταές ε, πήρε την ευθύνη, ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης και αυτό δείχνει ακόμη μια φορά πόσο βάρβαρη είναι η ιδεολογία του που συνίσταται σε μια πολιτική μορφή του Ισλάμ και απόρριψη του άλλου. Η ίδια μυσαλλοδοξία και βαρβαρότητα χτύπησε την περασμένη Παρασκευή στην Ιεμένη και τους χριστιανούς στο Πακιστάν στις 15 Μαρτίου. Προστά σε όλα αυτά πρέπει περισσότερο από κάθε άλλη φορά να επιμείνουμε στις αξίες μας, να καταπολεμήσουμε τον φανατισμό και την τρομοκρατία με τους εταίρους μας και κυρίως με την Τινησία. Υποστηρίξαμε τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας αυτής από την αρχή και δεν πρέπει να την εγκαταλείψουμε τώρα αυτή την κρίσιμη ώρα. Χρειάζεται μια διεθνής βοήθεια και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί υπάρχει Πάτη εκπρόσωπος σε όλες τις πτυχές της συνεργασίας μας ετέχθη, τάχθη υπέρ. Εξάλλου σε λίγο μια αντιπροσωπεία συναδέλφων που είναι τμήμα της αντιπροσωπείας μας με το που θα πάει στην Τινησία για να ανταλλάξει απόψεις με τους κοινοβουλευτικούς εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε Πρέντα. Ακολουθεί ο συνάδελφος Παντσέρη, μισή λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ επέστρεψα σήμερα το πρωί από την Τίνιδα, είχα κάποιες επίσημες επαφές και με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου που μου επιβεβαίωσε ότι βασικός στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης ήταν η Βουλή. Αντάλλαξα απόψεις με αρκετούς Τινησίους και κατάλαβα ότι η Τινησία θα έπρεπε, είναι ένα ιδανικό θέατρο για επιθέσεις τρομοκρατικές. Η χώρα αυτή που γέννησε την Αραβική Άνοιξη είναι και η χώρα που έχει κάνει τα περισσότερα βήματα στον τομέα της ε, ε, μετάβασης προς τη δημοκρατία. Έχει υιοθετήσει ένα σύγχρονο συνταγματικό χάρτη και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε με θετικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τινησία χτυπήθηκε γιατί η θετική κατάληξη της προσπάθειας που γίνεται εκεί θα ήταν σημείο αναφοράς ε, για ε, όλη την περιοχή. Θα ε, ήταν η απόδειξη, αν θέλετε, ότι μπορεί να υπάρξει δημοκρατικό μέλλον για τις αραβικές χώρες. Και αυτό για τους τρομοκράτες δεν είναι ανεκτό, γιατί έχουν σαν στόχο το χάος σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της χώρας. Η τρομοκρατία δεν είναι μόνο πρόβλημα της Τινησίας, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Οι επιθέσεις το Μουσείο Μπάρντο προκάλεσαν θύματα και ανάμεσα σε Ευρωπαίους επισκέπτες. Από τη μία αυξάνεται ο φόβος για τις επισκέψεις σε αυτές τις χώρες και από την άλλη υπάρχει μία μείωση της διεθνούς εικόνας της χώρας και καταλαβαίνετε τι συνέπειες ε, θα υπάρχουν από τη μείωση των εσόδων στον τομέα του τουρισμού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μην μιλάμε πολύ και θα πρέπει να βοηθήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο σήμερα. Η Ευρώπη έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει απέναντι στην την σε δύο τομείς. Καταρχάς, πολιτική στήριξη των, την, των θεσμών της δημοκρατίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα αντισώματα τα οποία θα αντιπαρατεθούν με τον Ισλαμικό κίνδυνο και από την άλλη, όπως είπε και η κυρία Μογκερίνη, θα πρέπει να βοηθήσουμε σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και οικονομικά άμεσα. Όπως βοηθήσαμε την Ουκρανία πρόσφατα στον τομέα των οικονομικών. Νομίζω ότι αυτό θα αποδείξει την επιτυχία της νέας πολιτικής γειτονίας της δυνατότητας που έχει η πολιτική αυτή να είναι ευέλικτη, να εντοπίζει τις προτεραιότητες. Εμείς οι σοσιαλιστές πιστεύουμε ότι η Τινησία συνιστά μία προτεραιότητα. Γνωρίζω την ευαισθησία σας κυρία Μογκερίνη. Θα ήθελα όμως να δεχθείτε το αίτημά μας και να υπάρξει πέρα από αυτά τα οποία είπατε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη συνάντηση του μηνός Μαΐου έτσι ώστε τέτοιου είδους συμβάντα να μην επαναληφθούν σε χώρες στις οποίες θέλουμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφε Παντσέρη. Ένα λεπτό τώρα ο συνάδελφος Τάνοκ παρακαλώ. Εκφράζω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια των θυμάτων για την επίθεση του Μπάρντο όπου σκοτώθηκαν 23 άτομα με, από επίθεση με αυτόματα κατά αθώων τουριστών και πολιτών. Η Ισλαμική οργάνωση ανέλαβε, το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη και είτε είναι αλήθεια αυτό είτε όχι, δείχνει αυτό την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι Ισλαμιστές τρομοκράτες κατά της Ευρώπης. Οι τρομοκράτες αυτοί δεν ενδιαφέρονται ποιον σκοτώνουν, μουσουλμάνους, χριστιανούς ή Εβραίους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καταστροφή όσων θεωρούν αντίπαλους του λεγόμενου χαλιφάτου των. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί άνθρωποι και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στις χώρες μας και οικονομικά και ως προς την ασφάλεια για να βοηθήσουμε την νεαρή δημοκρατία της Τινησίας. Ευχαριστώ συνάδελφε Τάνα. Δύο λεπτά Μάουρα Μπαραντιαράν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακριβώς όπως και στη συζήτηση για τη Λιβύη που έγινε σε προηγούμενη ολομέλεια για την αποσύνθεση αυτής της χώρας που ήδη έφτασε τώρα στην ε, την Ισία και δηλώθηκε στην ίδια αυτή συζήτηση για την κατάσταση στη Λιβύη και στο, τη Βόρεια Αφρική είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και η Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά αυτές οι προτεραιότητες ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά αντανακλώνται. Δύο τρίτα των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας στοχεύουν σε περιοχές ε, της Ανατολικής Ευρώπης με 12 εκατομμύρια κατοίκους ενώ στο Νότο με 22 εκατομμύρια, 22 εκατομμύρια πληθυσμό δεν δίνεται ίδια προτεραιότητα. Πρέπει εδώ να υπάρξει ισορροπία προτεραιοτήτων. Η κατάσταση νότια της Ευρώπης είναι πραγματικά οξύτατη και ακραία. Πρέπει κατεπηγόντως να αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας ώστε να εγγυάται με ισορροπημένο τρόπο την δέσμευση που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους γείτονές της. Στην περίπτωση της Τινησίας η επίθεση των τρομοκρατών την προηγούμενη εβδομάδα πέρα από την αναζήτηση αποσταθεροποίησης ήθελε να πλήξει τον πιο σημαντικό παραγωγικό τομέα, τον τουρισμό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι είναι η μόνη χώρα όπου πραγματικά η δημοκρατία έχει προχωρήσει. Πουθενάλλου δεν υπάρχει ε, μια κυβέρνηση που να έχει κερδίσει με τον ίδιο τρόπο τις εκλογές. Δεν υπάρχει σε, άλλο, ε, σε άλλη χώρα στο νότο της Ευρώπης ε, χώρα που να μην είναι ε, μια δικτατορία εκτός από την, την Και εδώ λοιπόν το Ισλαμικό κράτος θέλει να νικήσει αυτή την κυβέρνηση να ανατρέψει την κατάσταση. Πρέπει να δράσουμε με κάθε μέσο. Να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δάνεια, με χορηγίες, με κονδύλια που θα διατεθούν. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ούτε μία άλλη αιστεία αστάθειας στα νότια σύνορα της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ συνάδελφε Μαουρα Μπαραντιαράν. Για μισή λεπτό κόσο περνούει παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Μογερίνη που ήρθατε και πάλι στην Ολομέλεια να καταδικάσουμε και να εκφράσουμε τη θλίψη μας για τις πολλές αυτές επιθέσεις εξ ονόματος της ε, θρησκευτικής ε, τρομοκρατίας ε, και των εξτρεμιστών. Υπήρξαν τέτοιες απόπειρες και δεν τους δώσαμε πολύ, μεγάλη σημασία. Στην τοποθέτησή σας είπατε εκπρόσωπε, είπατε σε σχέση με τη Λιβύη για την ίδια κατάσταση και έχει δίκιο αυτό διότι δεν είναι δυνατόν η τρομοκρατία ανά χώρα να καταπολεμάται Πρέπει εδώ λοιπόν σε σχέση με τη Μέση Ανατολή πραγματικά να δούμε ότι η υποστήριξη δικτατόρων δημιούργησε τέρατα όπως το Ισλαμικό κράτος και πρέπει να το πούμε αυτό. Και έτσι λοιπόν πρέπει η πολιτική αυτή της ανάμειξης, οι, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπάθησαν να ε, βοηθήσουν τις μοναρχίες και τους δικτάτορες της Μέσης Ανατολής και διάφορες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν αυτή την Το Ισλαμικό κράτος πολύ καλά χρηματοδοτείται σήμερα και είναι κάθε φορά όλο και πιο ισχυρό στη Μεσόγειο, διότι πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφεραν να καταστραφούν οι δομές του κοσμικού κράτους. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον ρόλο των περιφερειακών εμπλεκόμενων. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον ρόλο των πολυεθνικών θεσμικών οργάνων. Και έτσι λοιπόν οι ε, αυτοκρατορικές περιπέτειες που ακολουθούν ακολουθήθηκαν βλέπουμε ότι οδήγησαν σε αυτά τα ικτρά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Λοχ Μπίλερ παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ πρόεδρε η επίθεση στο Μουσείο Μπαρντό στην την, την κόστισε, ε, είχε 22 θύματα και το Ισλαμικό κράτος δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνο. Εσείς κυρία Μογκερίνη αμέσως μετά την, ε, το πλήγμα αυτό υποστηρίξατε την κυβέρνηση της Τινησίας και όχι μόνο με μέτρα ασφάλειας αλλά και την, για την οικονομική και δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας και το κάνατε αυτό και σήμερα διεξοδικά αναφέρατε τα σχετικά. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να εκφράσει την αλληλεγγύη της με την Τινησία σε σχέση με αυτές τις δύσκολες χρονικές στιγμές. Στα λόγια μας όμως πρέπει να ακολουθούν πράξεις και να δώσουμε τα επαρκή κονδύλια που θα διαθέσουμε ώστε να υποστηριχτεί η ε, χώρα αυτή και η υποστήριξη πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτό το πλήγμα δεν θα οδηγήσει σε μια οπισθοδρόμηση στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Τινησία ώστε η Τινησία να συνεχίσει να είναι ένα οικονομικό και δημοκρατικό πρότυπο Χιλιάδες Τινήσοι κατέβηκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν με αυτές τις ε, διαδηλώσεις όμως ε, εκφράστηκε και ε, με τροποποιημένο τρόπο η υποστήριξη για την επανάσταση που έλαβε χώρα στην Τινησία. Είπαν δεν φοβόμαστε πια, δεν φοβόμαστε σήμερα την τρομοκρατία. Μια και υπάρχει παγκόσμια οικουμενική απειλή από τζιχαντιστές, αυτό δεν πρέπει να είναι μόνο ένα κύριο μήνυμα για την Τινησία, αλλά για το σύνολο της περιφέρειας των περιοχών αυτών του κόσμου. Δεν φοβόμαστε την τρομοκρατία όμως αυτό να είναι και μια, ένας κόδωνας κινδύνου που κρούεται έναντι βιαστικών συμπερασμάτων και δράσεων. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους τινήσιους ώστε μέτρα για την προστασία από την τρομοκρατία να συνάδουν με την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών και θεμελιωδών αξιών. Ιδιαίτερα υπέρ των, ε, θεσμικών οργάνων του κράτους δικαίου και ιδιαίτερα όσον αφορά το κοινωνικό βήμα, κοινωνικό φόρουμ, το ότι διεξάγεται αυτό είναι μια χειροπιαστή έκφραση αλληλεγγύης προς τους τινήσιους και την κοινωνία τους. Ευχαριστούμε κυρία Λόχμπιλερ. Δύο λεπτά, συνάδελφε Καστάλτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Γιατί η τραγωδία αυτή χτύπησε την Τινησία. Τους τελευταίους μήνες πήγα τρεις φορές στην Τίνιδα για τις εκλογές στην χώρα όπου η Αραβική Άνοιξη πραγματικά δημιούργησε πολύ θετικά αποτελέσματα. Σήμερα βλέπω ότι οι φρικτές εικόνες του μουσείου δεν θα σβήσουν τις ωραίες εικόνες που έχω κρατήσει από τις επισκέψεις μου. Για μια ακόμη φορά λοιπόν λέγω α, εκ μέρους των Τινησίων Σούκραν. Ευχαριστούμε που βοηθάτε για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και στα εκλογικά γραφεία και ε, στις δημόσιες υπηρεσίες ε, και στα μουσεία, σε αυτό το εξαιρετικό μουσείο Μπάρτο και στα μοσαϊκά που ε, είναι μάρτυρες της σχέσης της στενής ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη έχει ανάγκη τον τουρισμό ή την Ισία για να βοηθήσει ε, την χώρα να βγει από την φτώχεια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες θέλουν ακριβώς με τον τρόμο να δείξουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο Ισλάμ και τη Δημοκρατία. Και δυστυχώς αυτό το έχουν και άλλοι σαν συμφέρον. Υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ε, ε, στο σοκ των πολιτισμών, στο σοκ των θρησκειών ο βασιλιάς της Ιορδανίας είπε ότι οι μουσουλμάνοι στον κόσμο δεν θα επιτρέψουν στους τρομοκράτες να εκμεταλλευτούν την πίστη τους για λόγους βαρβαρότητας. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ακόμα περισσότερες προσπάθειες. Μόνο αν συνεργαστούμε στενά στον οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό τομέα θα μπορέσουμε να νικήσουμε ε, την, ε, τον πολιτισμό της βίας ε, με την δύναμη του πολιτισμού. Είμαστε όλοι την ίση. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο. Ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ την κυρία Μογκερίνη. Φυσικά και εμείς συμμεριζόμαστε τα συλληπιτήρια. Πολλοί από τους νεκρούς είναι συμπατριώτες μας, αλλά το ίσις δεν κατεπολωμάται από προσευχές είτε στην αραβική είτε στη λατινική γλώσσα. Πρέπει να δώσουμε μέσα στρατιωτικά, μέσα κατασκοπίας, συλλογής πληροφοριών και όχι μόνο να στέλνουμε κάποιους, ε, κάποιους ε, διπλωμάτες και γραφειοκράτες που κάνουν διακοπές σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Πρέπει να σφραγίσουμε τα σύνορα με τη Λιβύη σαν παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν τα κροκοδίλια δάκρυα κάποιων κυβερνώντων που δεν έκαναν τίποτα μέχρι τώρα για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό των τρομοκρατών αλλά είναι πρώτοι στις κηδείες να κλαίνε μπροστά στις κάμερες για τα θύματα. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον κίνδυνο αυτό και να βοηθήσουμε τη φτωχή αυτή χώρα. Ας πάμε όλοι για διακοπές στην Τινησία πια. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Μποκέσιο για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση και πάλι τώρα η Επίτροπος κυρία Μογκερίνη. Ε, Θα απαντήσω προς τον κύριο Μποργκέτσιο να πω ότι το θέμα του ελέγχου ανάμεσα στην Τινησία και τη Λιβύη είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τινησίας μια μέρα πριν από την επίθεση στον Πάρντο. Αυτός είπε ότι η Τινησία δεν έχει καμία πρόθεση να σφραγίσει τα σύνορα με την Λιβύη. Εγώ έχω συνηθίσει να σέβομαι αυτά τα οποία επιθυμεί μια χώρα. Ιδιαίτερα όταν λέμε ότι είναι μία από τις χώρες οι οποίες με επιτυχία ακολουθούν το δρόμο για τη δημοκρατία. Βάσει της σχέσης μας με την Τινίδα είναι ο σεβασμός της αποφάσεις της Τίνιδας και στις επιλογές της Τίνιδας. Είναι σαφές ότι δεν έχουμε να κάνουμε με σύγκρουση ανάμεσα σε πολιτισμούς και σύγκρουση ανάμεσα σε θρησκείες. Νομίζω ότι όλοι οι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, άφεοι, την ίση οι Ευρωπαίοι καταδικάζουμε τις επιθέσεις αυτές. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια διαφορά ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο. Υπάρχει μια κοινή προσπάθεια, μια προσπάθεια δύσκολη, μια προσπάθεια συγκεκριμένη όμως, έτσι ώστε από κοινού και στις δύο πλευρές της Μεσογειακής Λεκάνης να κάνουμε αυτά που πρέπει ενάντια στην τρομοκρατία. Σε ένα κλίμα ασφάλειας, με μέτρα ασφάλειας την... πρέπει να τα πάρουμε τα μέτρα αυτά, αλλά θα νικήσουμε μόνο αν μπορέσουμε να επενδύσουμε στις νέες γενιές, προσφέροντας θέσεις εργασίας, προσφέροντας θέσεις στην κοινωνία, προσφέροντας αξιοπρέπεια, γιατί αυτό ζητούν οι νέοι της Τινησίας ε, με την επανάστασή τους πριν μερικά χρόνια. Πρέπει λοιπόν εμείς ε, να υποστηρίξουμε με σεβασμό την πορεία της Τινησίας με όλα μας τα μέσα, σεβόμενοι όμως την αξιοπρέπεια της χώρας αυτής και του λαού της. Για κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα, το πρώτο αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας. Αυτά είναι ένα θέμα από τα θέματα που συζητήσαμε με τους Τινήσιους μία μέρα πριν από την απόπειρα την τρομοκρατική. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και στη Βαρκελόνη στις 13 Απριλίου και θα τα συζητήσουμε επίσης και με τους ανατολικούς μας εταίρους το μήνα Μάιο. Η αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας και για μας και για τους εταίρους μας είναι ένα καταπληκτικό μέσο αν <clears throat> το αντιληφθούμε σαν γραφειοκρατική διαδικασία δεν θα αποδώσει. Αλλά όπως είπα με αμοιβαίο σεβασμό θα μπορέσουμε εμείς να βρούμε τα μέσα ε, τα οποία θα μας επιτρέψουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της σταθεροποίησης της περιοχής, ε, της τρομοκρατίας, ε, της καταπολέμησης του έφραστου χαρακτήρα των κρατικών δομών Βλέπουμε τι γίνεται στη Λιβύη. Ε, τα θύματα είναι όλα δίκαια και ισότιμα. Ε, ξέρετε ότι ε, δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα στα θύματα. Όλα τα θύματα είναι σημαντικά και θα ήθελα να αναφερθώ και σε θύματα σε άλλες περιοχές του κόσμου όπως η Αλγερία, όπως την Ιεμένη Ξέρετε ότι γίνεται στην Ιεμένη σήμερα. Θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και θα πρέπει επίσης να προσέξουμε έτσι ώστε οι περιφερειακές κρίσεις να μην διαδίδονται. Και γι' αυτό εδώ έρχομαι ε, σε αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις όχι μονομερείς αλλά πολυμερείς. Η έκκληση αυτή είναι και δική μου έκκληση. Είναι μια έκκληση που κάνω καθημερινά και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και σε επίπεδο Αραβικού Συνδέσμου. Έχει μεγάλη σημασία όλοι οι εμπλεκόμενοι στην περιοχή να δράσουν με ευθύνη, με αίσθημα υπευθυνότητας και όχι μόνο για τη Λιβύη αλλά και για την Ιεμένη. Έχουμε ένα πλαίσιο πολυμερών σχέσεων και μέσα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δράσουμε, να δράσουμε σωστά, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις και αυτό δείχνει ότι ένας από τους τρόπους επίλυσης μιας κρίσης, ο πιο εύκολος είναι το να δημιουργήσει μια νέα κρίση. Πρέπει να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο κυρίως στη Λιβύη θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε μελλοντικές κρίσεις και να περιορίσουμε τις τρομοκρατικές δράσεις στην περιοχή. Μία τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την κατανομή των πιστώσεων. Κάποιοι από σας αναφερθήκατε σε μία άνεση κατανομή δύο τρίτα για την Ανατολή και ένα τρίτο για τον Νότο. Είναι ένας κανόνας που δεν είναι καταγεγραμμένος. Πράγματι τα δύο τρίτα δίδονται στον Νότο και το ένα τρίτο στην Ανατολή. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να τα διευκρινίσουμε γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα δημιουργηθούν συγχύσεις. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μογκερίνη, κυρία Επίτροπε Μογκερίνη. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτού του θέματος.